Good morning. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης σήμερα. Έχουμε προσκαλέσει τον καθηγητά Στικλίτ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο και τον καθηγητή Οκάμπου πρώην Υπουργό τη ε, Κολομβίας και τώρα καθηγητή από το Κολούμπια και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Σήμερα είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να καλωσορίσω τον καθηγητή Στίγκλιτς, Νόμπελ Οικονομικών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε για την προθυμία σας σας προσκαλέσαμε ως πρώην εμπειρογνώμονα της ε, εκταστική Επιτροπής ε, για το σκάνδαλο Panama Papers και θέλουμε να έχουμε διάλογο μαζί σας βάσει της ε, πείρας που διαθέτετε στα πλαίσια αυτής της Εκθεστικής Επιτροπής. Σας έχουμε στείλει ένα κατάλογο με ερωτήσεις Και πραγματικά είναι τιμή μα που κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου βρήκατε χρόνο για να απαντήσετε. Οι απαντήσει σα έχουν μοιραστεί στα μέλη της Επιτροπής μας. Μετά τα εισαγωγικά σα σχόλια, εάν μπορείτε σε 10 λεπτά, θα δώσω το λόγο σε ένα γύρο απαντήσεων από τους συναδέλφους. Έχουμε 14 γλώσσες σε διερμηνία σήμερα. Οι ερωτήσεις θα τεθούν σε χρονοθυρίδες του πεντάλεπτου, ίσως να περιοριστούμε στα τρία λεπτά σήμερα. Ερώτηση ένα λεπτό και ο υπόλοιπος χρόνος απάντηση. Καθηγητά Στίγλιτς, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Well, thank you very much for this opportunity to... Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα ενώπιον σας. Νομίζω πως το αντικείμενο της Επιτροπής σας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η φορολογική παράδειση που ήρθαν στην επιφάνεια μετά τη, τα Panama Papers είχαν ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, καταστροφικές επιπτώσεις για την κοινωνία μας, την παγκόσμια κοινωνία. Η φορολογική παράδειση αυτή είναι κέντρα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, ε, υποστηρίζουν και στηρίζουν τη διαφθορά, βοηθούν στο ξέπλυμα χρήματος, ε, είναι κέντρα διαφόρων τέτοιων δραστηριοτήτων και Όταν ήρθαν λοιπόν στο προσκήνιο τα Panama Papers, μας βοήθησαν να συνειδητοποιήσουμε την κλίμακα στην οποία ε, γίνονται όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ε, δραστηριότητες, σκοτεινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, όμως τα Panama Papers κατάφεραν να ρίξουν φως σε ό,τι συνέβαινε. Και θα ήθελα να τονίσω ότι το 80% των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα και που περιγράφουν τα Panama Papers δεν έλαβε χώρο στον Παναμά. Αυτό τονίζει τον καθολικό οικουμενικό χαρακτήρα του προβλήματος. Το σκάνδαλο αυτό ήρθε στην επιφάνεια εν μέρη επειδή στην αγγλική γλώσσα είχε έτσι ένα πιασάρικο όνομα. Panama Papers, όπως Leaks. Και αυτή λοιπόν η ονομασία έτσι βοήθησε στο να γίνουν πιο γνωστά. Στο επίκεντρο του σκανδάλου ήταν μια νομική εταιρεία του Παναμά η οποία είχε αναλάβει όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες. Ε, άνοιξε λοιπόν το κουτί της Πανδώρας και δημοσιεύτηκαν πάρα πολλά έγγραφα. Και θυμηθείτε πως ε, αυτή ήταν μόνο μία εταιρεία. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες τέτοιες εταιρείες στον Παναμά και η συγκεκριμένη είναι από τις μικρότερες. Όπως μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε, όταν μία τόσο μικρή εταιρεία βοήθησε να έρθουν στο φως ε, τόσο πολλά σκάνδαλα, αλλά φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες που είναι μεγαλύτερες. Και γενικά τι συμβαίνει σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Και θα ήθελα να πω σε όσους δεν είχαν την ευκαιρία να κοιτάξουν τις γραπτές μου απαντήσεις, ότι μετά ε, τα Panama Papers, όταν λοιπόν ήρθαν αυτά στη δημοσιότητα, ε, ο Παναμάς ε, θεώρησε πως έχει υποστεί ε, μεγάλο πλήγμα ως χώρα. Η φήμη έχει πληγεί και μάλιστα μετά το παρελθόν του Νουριέγκα και των ναρκωτικών θεώρησε η κυβέρνηση του Παναμά ότι πρέπει να επανορθώσει το κακό που έχει γίνει. Εγώ ήλπιζα να ήθελαν πολύ περισσότερο από αυτό, όχι μόνο δηλαδή να αποκαταστήσουν την ε, φήμη τους, αλλά να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Έτσι λοιπόν ε, προσπάθησαν να με πείσουν να γίνω μέλος μιας επιτροπής μαζί με τον Μαρκ Πάιτ, έναν έγκριτο νομικό, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές εκστρατείες ε, κατά της διαφθοράς τα τελευταία 25 χρόνια. Μας κάλεσαν λοιπόν να συμμετέχουμε σε αυτή την επιτροπή και ένας από τους λόγους που δέχτηκα ήταν ότι πίστευα πως η δουλειά μας θα αποτελούσε υπόδειγμα για τη συνέχεια. Είχαμε δηλαδή το παράδειγμα μιας χώρας που ήθελε να κάνει μεταρρυθμίσεις, που ήθελε να δώσει το καλό παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Και να σας πω πως ε, ήθελα ο Παναμάς να αποτελέσει υπόδειγμα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν και αυτές φορολογικούς παραδείσους, διάφορες πολιτείες, στο Delaware, στην Εβάδα και σε άλλες. Ήλπιζα λοιπόν, μελετώντας την περίπτωση μίας μικρής χώρας, να καταφέρουμε να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο στη συνέχεια θα ε, μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Στην αρχή των ε, διαπραγματεύσεών μας είπαμε στην κυβέρνηση του Παναμά πως θέλαμε κάποιες διασφαλίσεις ότι η έκθεσή μας θα χαρακτηριζόταν από διαφάνεια και πώς θα δημοσιευόταν αφού η κυβέρνηση του Παναμά είχε αρκετό χρόνο για να επεξεργαστεί μία απάντηση. Περιμέναμε εβδομάδες, εβδομάδες επί εβδομάδων και η κυβέρνηση δεν μας έδωσε αυτές τις διασφαλίσεις και στο τέλος ε, μάθαμε πως ε, δεν υπήρχαν τέτοιες διασφαλίσεις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε πως ε, ήταν καθήκον μας να παρετηθούμε. Όμως νομίζω πως αυτόν τον καιρό που εργαστήκαμε στην Επιτροπή αυτή βρήκαμε αρκετά στοιχεία ικανά για να αποτελέσουν μέρος μιας έκθεσης η οποία θα συνόψιζε τα όσα καταφέραμε να βρούμε. Και να αποκρισταλώσω κάποιες θέσεις μας για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της έκθεσής μας, η σκιώδης οικονομία δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα ήθελα να κάνω μια σύντομη περιγραφή των κεντρικών θεμάτων της έκθεσής μας. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αυτή η φορολογική παράδειση αποτελούν το σκοτεινό μέρος, τη σκοτεινή πλευρά της παγκοσμιοποίησης. κρύβονται χρήματα, εξαφανίζονται χρήματα. Είτε αυτά έχουν προέλθει από φοροαποφυγή, από ξέπλυμα, από παράνομες δραστηριότητες και όλο αυτό υπονομεύει την ομαλή λειτουργία ε, της παγκόσμιας κοινωνίας. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε πριν τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ, στις εκλογές δηλαδή της περασμένης εβδομάδας. Και νομίζω πως αν δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες μας ότι μπορούμε να αμβλύνουμε τις ε, άσχημες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, οι εξελίξεις αυτές ολοένα και θα αυξάνονται. Θα έχουμε πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις. Σίγουρα η παγκοσμιοποίηση έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, είναι σε γενικές γραμμές κάτι θετικό, πρέπει όμως να μην παραγνωρίζουμε τις δυσάρεστες συνέπειες, τη σκοτεινή της πλευρά. Και κάτι το οποίο επίσης τονίζουμε στην έκθεση, είναι πως χρειάζεται μία ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για τους φορολογικούς παραδείσους. Εάν υπάρχει έστω και ένα μέρος σε αυτόν τον πλανήτη που να λειτουργεί ως φορολογικός παράδεισος, τότε θα προσελκύσει όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Τότε θα κρύβονται όλοι εκεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μία ολοκληρωμένη περιεκτική προσέγγιση με μηδενική ανοχή για τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό σημαίνει βεβαίως πως ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό παγκόσμια και συνολικά. Και θεωρώ επίσης πως ε, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, είναι ένα αρκετά περίπλοκο και πολύπλοκο ζήτημα. Όταν όμως αντιμετωπίσαμε ε, πάλι παγκόσμια το φαινόμενο της τρομοκρατίας, καταφέραμε πολλά. Καταφέραμε να εντοπίσουμε προς τα που πήγαιναν τα χρήματα που στήριζαν ε, την ε, τρομοκρατία. Δεν έχουμε καταφέρει όμως να το κάνουμε ακόμα ούτε για την ομοιοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ούτε για την ε, αποφυγή και φοροδιαφυγή. Και αυτό μου θυμίζει μία ομιλία που είχα κάποτε, που είχε ακριβώς αυτό το θέμα με κάλεσα να κάνω μια διάλεξη ακριβώς σε έναν από αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους για, το, για τις συνέπειες που έχουν οι δραστηριότητες αυτές στην παγκόσμια οικονομία. Και είχα την εντύπωση ότι τους άρεσε πάρα πολύ η ομιλία μου, πως ήταν καθαρτική για κοινούς, έτσι ώστε να συνεχίσουν με καθαρή συνείδηση τις παράνομες δραστηριότητες τους. Και μάλιστα θυμάμαι πως με πλησίασε ένας ε, τραπεζίτης και μου είπε πως ε, δεν καταλαβαίνετε το πώς δουλεύουμε εδώ. Ε, δεν κάνουμε αυτά που είπατε, δεν ασχολούμαστε με ναρκοδολάρια, δεν συμμετέχουμε σε χρηματισμού, σε διαφθορά. Όχι, όχι, εμείς μόνο φοροδιαφεύγουμε. Μόνο με αυτό ασχολούμαστε. Και τους ρώτησα λοιπόν πώς το ξέρετε. Ε, μα τους ρωτήσαμε ξέρετε μου απάντησαν. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα εδώ. Χρειάζεται συνολική καθολική αντιμετώπιση και πιστεύω πως ε, η Ευρώπη μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ σημαντικά, να κάνει τη διαφορά. και κάτι που υπογραμμίζουμε στην έκθεση αυτή είναι ότι σε αυτές τις δραστηριότητες δεν συμμετέχουν μόνο εξωχώριες εταιρείε, αλλά ε, και εντός συνόρων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις και των Ηνωμένων Πολιτείων και των Ευρωπαϊκών χωρών να το καταπολεμήσουν. Η περίπτωση του Panama Paper ήταν πιστεύω η αρχή το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αντιδράσει, έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα της, ε, του κύριου, των κύριων δικαιούχων και ελπίζω το έργο που άρχισε η προηγούμενη κυβέρνηση να συνεχίσει και η επόμενη, διότι ως γνωστόν ο επόμενος πρόεδρός μας είναι διαβόητος για θέματα φοροδιαφυγής. Και όταν μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος φοροδιαφεύγει ή φοροαποφεύγει, μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στο έργο μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ακόμα σημαντικότερο εξαιτίας αυτού η Ευρώπη να αναλάβει τα ενία αυτής της εκστρατείας. Κάτι άλλο που τονίζουμε στην έκθεσή μας είναι ότι το φαινόμενο αυτό ξεπερνά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, εστιάζουμε βέβαια σε τράπεζες, οι οποίες σίγουρα έχουν διαδραματίσει ένα πολύ άσχημο ρόλο σε όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες. Και μιλάμε για μεγάλα ποσά εδώ. Όμως πιστεύω πως οι τράπεζες έχουν καταφέρει να κάνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, ακριβώς επειδή είχε δοθεί τόσο μεγάλη προσοχή σε αυτές. Αναγκάστηκαν λοιπόν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις κατηγορίες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν. Όμως πέρα από τον ε, τραπεζικό τομέα υπάρχει ένας ε, τεράστιος κλάδος, ένα τεράστιος χώρος μάλλον, με πολλού κλάδου που ε, συμμετέχει σε αυτέ τι δραστηριότητε, ε, νομικές ένα παράδειγμα μόνο και από αυτές μάλιστα ήρθε στην επιφάνεια όλο αυτό το φαινόμενο. Και προτείνουμε στην έκθεσή μας αυστηρά μέτρα αντιμετώπισης ε, για αυτές τις εταιρείε. Και κάτι άλλο. Η έκθεσή μας επίσης ε, αναφέρει πως ε, πολλές χώρες θα υπογράψουν συμφωνίες περί διαφάνειας, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Θα υπογράψουν συμφωνίες για πολλά μέτρα και αφού υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες μπορούν όλοι να κοιμούνται ήσυχοι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί το σημαντικό, πρωταρχική σημασία είναι η εφαρμογή των νόμων, η εφαρμογή μιας συμφωνίας, διότι όλοι ξέρουν ότι μπορείς απλά να υπογράψεις και να μην κάνεις τίποτα. Και μπορείτε να φανταστείτε πως η δικαστική εξουσία σε πολλέ χώρες δεν είναι ακριβώς σε θέση η πρόθυμη να εφαρμόσει όλε αυτές τις συμφωνίες. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ διεθνή προσέγγιση. Διότι δεν έχει σημασία μία συμφωνία, σημασία έχει η εφαρμογή της. Η έκθεσή μας επίσης περιέχει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις ε, συνέπειες του φαινομένου και με τις αρχές που διέπουν τη σκιώδη οικονομία και μια αντιμετώπιση αυτής. Πιστεύω πως αν έπρεπε να απομονώσουμε ένα στοιχείο το οποίο μπορεί από μόνο του να κάνει τη διαφορά, αυτό θα ήταν η πραγματική κυριότητα μιας εταιρείας. Γιατί ακριβώς όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις σκιώδεις δραστηριότητες αποτελούν έναν κρίκο μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας. Μία ας πούμε μυστική εταιρεία αλφα είναι ιδιοκτήτρια μια άλλη εταιρεία Β, που με τη σειρά τη είναι ιδιοκτήτρια μια εταιρεία Γ. Και έτσι λοιπόν δυσκολεύει πολύ το έργο του να εντοπίσει τον πραγματικό δικαιούχο. Αυτό είναι ένας ιστός ο οποίος είναι τόσο πυκνός που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των αρχών για να εντοπίσουν τον τελικό πραγματικό δικαιούχο. Χρειάζεται λοιπόν καταρχάς ένα μητρό αυτών των ε, πραγματικών δικαιούχων, όχι αυτών των ε, εταιριών, των ψεύτικων εταιριών, ονόματα. Αυτό είναι η της σημασίας. Και αυτό το μητρό πρέπει να είναι ανοιχτό, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο οι αρχές επιβολής νόμου, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να αναζητήσουν το ποιος κάνει τι. Όμως αυτός ο περίπλοκος ιστός δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούν μόνο οι πολυεθνικές. Υπάρχουν και ε, πολλές θηγατρικές εταιρείες. Αλλά τι γίνεται εκεί. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν αυτό τον ιστό. Γιατί, πολύ απλή απάντηση, για να μην πληρώσουν φόρους. Για παράδειγμα, προσπαθούν να αποφύγουν την ανάληψη ευθυνών, προσπαθούν να αποφύγουν τις μηνύσεις. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν γίνονται με διαφάνεια, δεν γίνονται δημόσια. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο όσοι ασκούν παράνομη δραστηριότητα, που χρησιμοποιούν αυτόν τον περίπλοκο ιστό, είναι και πολύ μεγάλες, αξιοσέβαστες εταιρείε, καθόλου νόμιμέ κατά τα άλλα. Αλλά ας δούμε και το φαινόμενο αυτό στο κοινικότερο πλαίσιο και ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Το θέμα είναι πως πρέπει να αποκαλύψουμε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συνεχίσουν αυτό το σκοτεινό τους έργο, το να υπονομεύουν δηλαδή ε, την παγκόσμια κοινότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Στίκλιτς για αυτήν την ενδιαφέρουσα και ανοιχτή εισαγωγή. Τώρα κυρίσω την έναρξη της συζήτησης με τα μέλη της Επιτροπής ΠΑΝΑ. Θα αρχίσω με τους δύο συνεισηγητές μας. Γέπε Κόφορτ και Πέτερ Γέτσεκ. Γέπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Τζο για αυτή την άρεστη παρουσίαση. Έχω τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα στην εγγραφή απάντησή σας είπατε πως η μυστικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί επάκτια και παράκτια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή βρεχή πρόθεσμα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως διεθνής κοινότητα. Υπάρχει ανάγκη σύγκλησης μιας ε, Διεθνού συνόδου για το ζήτημα της μυστικότητα. Έχουμε συνόδους για την κλιματική αλλαγή και τέτοια θέματα. Δεύτερον, σε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζητήσαμε να συσταθεί ένα παγκόσμιο μητρό των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων εταιριών. Αυτή είναι μια εφικτή ιδέα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ποιο θεσμό θα μπορούσε να το παράσχει. Τρίτον, μιλήσατε για κυρώσεις και συνέπειες για αυτούς που προβαίνουν σε φόρο διαφυγή και τα λοιπά, για νομικές εταιρείες, διαχειριστές. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να τους πάρουμε τις άδειες άσκηση επαγγέλματος. Τι είδους κυρώσεις είναι αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καθηγητά Στίγλιτς. πιστεύω πως η ιδέα μιας παγκόσμιας συνόδου είναι πολύ καλή. Και πιστεύω πως το ζήτημα που θέσατε είναι πως όντως πρόκειται για ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα. Και η εργασία του Ζουκμαν έδειξε παραδείγματο χάρη πως ο παγκόσμιος πλούτος διαφεύγει της φορολογίας και της δήλωσης. Τονίζω λοιπόν πως το πρόβλημα είναι χειρότερο στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη φορολογία, όχι την διαφθορά. Για τους εξής λόγους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η φορολογία βασίζεται στην ηθαγένεια. Όταν ένας Αμερικανός πολίτης λοιπόν δηλώνει τα εισοδήματά του όπου και αν τα επιτυγχάνει. Ακόμη και αν το κάνει σε κάποια νησιά. Στα νησιά Καϊμάν Γι' αυτό και καταρχάς το να πάει κανείς στις νήσους Καϊμάν δεν τον προστατεύει καταρχάς από την υποχρέωση του να δηλώσει το εισόδημά του. Εάν συστήσει μια εικονική εταιρεία μπορεί να αποφύγει την δήλωσή της μόνο εάν η αμερικανική συγκυριότητα είναι μειοψηφική. Εάν η πλειοψηφική συμμετοχή είναι ευρωπαϊκή, τότε υπάρχει υποβοήθηση της αμερικανικής πλευράς να κρυφτεί πίσω από το απόρριτο. Αλλά οι περισσότερε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η φορολογία βασίζεται στον τόπο εγκατάσταση, δηλαδή όπου οι άνθρωποι κερδίζουν το εισόδημά τους. Γι' αυτό και η προσέγγιση δεν είναι τόσο παγκόσμια όσον αφορά τη φορολογία. Γι' αυτό και η χρήση υπεράκτιων κέντρων ειδικότερα είναι πιο προβληματική στην περίπτωση της Ευρώπης. Και γι' αυτό είναι και πιο σημαντικό για την Ευρώπη από ό,τι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω όμως πως μια παγκόσμια σύνοδος θα μπορούσε να επιστήσει την προσοχή στο πρόβλημα αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Συνομίλησα με κάποιες άλλους φορολογικούς παραδείσους και τουλάχιστον ο ένας μου είπε πως δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συναλλαγές. Θα θέλαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά σε τι θα μας ωφελούσε αν ήμασταν καλύτεροι και τα χρήματα πήγαιναν κάπου αλλού. Είπαν λοιπόν πως θέλουν να είναι καλύτεροι πολίτες αν όλοι οι άλλοι είναι επίσης καλύτεροι. εάν σε μια παγκόσμια σύνοδο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέοι παγκόσμιοι κανόνες, τότε αυτή η δικαιολογία δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πλέον. Με ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να απευθυνθεί κανείς στις χώρες που υπονομεύουν τους παγκόσμιους κανόνες αυτούς. Γι' αυτό και πιστεύω πως μια παγκόσμια σύνοδος θα μπορούσε να θεσπίσει τέτοιους κανόνες και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, πιστεύω πως δεν υπάρχει κανένας λόγος κάθε επιμέρους χώρα να μην μπορεί να αποκαλύψει την πραγματική κυριότητα όλων των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στις χώρες αυτές. Αυτό ίσως ήταν ένας τέτοιος κανόνας που θα μπορούσε να θεσπιστεί. Στον Παναμά Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις καταχωρημένες και θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο, ο πραγματικός, ποια είναι η πραγματική κυριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τι κάνουν, γιατί υπάρχουν, αν επιτυγχάνουν εισοδήματα και ένα μέρος των θεμάτων που συζητούμε αναφέρονται στην αύξηση των απαιτήσεων απέναντι σε αυτές, δηλαδή να αναφέρουν τι κάνουν κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρές επιχειρήσεις και να ασχοληθούμε με αυτές που όντως υπάρχουν και να δούμε τι, σημαίνει, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στις επιχειρήσεις αυτές. Αυτό πιστεύω πως είναι εντελώς εφικτό. Τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν ανά τον κόσμο υπό την ευρεία έννοια για τα οποία κάθε χώρα θα έπρεπε να θεσπίσει ένα μητρό, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Και τέλος, όσον αφορά τις κυρώσεις, πιστεύω ένα από τα πράγματα που προτείνουμε είναι πολύ αυστηρές κυρώσεις κατά χωρών και εταιριών που δεν πληρούν αυτά που περιγράψαμε, συμπεριλαμβανομένου των περιπτώσεων που οι εταιρείε θα χάνουν την άδεια λειτουργία τους, λειτουργίας τους. Όσον αφορά τις χώρες, χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες διαφάνειας, θα πρέπει να αποκόπτονται αποτελεσματικά. Δηλαδή θα πρέπει να είναι παράνομο για τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβαίνουν σε συναλλαγές με χώρες η δικαιοδοσία των οποίων δεν πληρεί το διεθνέ δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο Πίτερ Γέτσεκ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε που είστε εδώ κύριε Στίγλιτς. Κάπου είπατε ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση, διεθνή ενίσχυση στις απαιτήσει. Και φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει τώρα από την Ένωση και θα μας έρθει και ο Ντόναλτ Τραμπ. Στο City του Λονδίνου, στις Βρετανικές Παρθένες νήσους, Και όταν άκουσα τι αναγγελίε του Αμερικανού Προέδρου, του νεοκλεγέντο Αμερικανού Προέδρου για τη νέα φορολογική του πολιτική και το πώ θα ξανακάνει μεγάλη την Αμερική, ακούσαμε ήδη ότι κάποιε εταιρείε φεύγουν ε, εκτό ε, ω φορολογική μανούβρα κιόλα. Αυτό σημαίνει ότι τα μετρητά, εφόσον επιστρέφουν για να φορολογηθούν στη χώρα, έχουν και 10% έκπτωση στις εταιρείε αυτές. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες φοροδιαφυγής και φοροαπάτης. Ευχαριστούμε πολύ, καθηγητά Στίκλιτ. Πολύ χοντρικά. Νομίζω το πρώτο θέμα που θέσατε για τη φοροδιαφυγή και την ε, φοροαποφυγή στο σύνδεο του Λονδίνου, στις Βρετανικές Παρθένους νήσους. Το τι προσπάθειες αποφυγής υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν νομοθεσίες, οι οποίες, νομοθετικά μέτρα, τα οποία δεν συνάδουν με αυτό που θα έλεγα εγώ χρηστά πρότυπα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως πρέπει να αναλάβει δράση αποφασιστικά και εσωτερικός δεν θα πρέπει να επιτρέπονται κάποια πράγματα. Σε κάθε μια από τις χώρες μέλη της και διεθνώς. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ και διάκριση μεταξύ ΕΠΑ και Παναμά. Ίσως από την οπτική γωνία της ε, Βαλτικής να μοιάζει δύσκολο αυτό, αλλά έτσι είναι. Εάν υπάρχουν ε, λιμένες απορρίτου εντός των ΗΠΑ, παραμένει πρόβλημα αυτό. Ξέρουμε ότι ε, το Υπουργείο Οικονομικών των Πολιτειών γνώριζε κάποια πράγματα για τον Παναμά. Ξέρουμε λοιπόν πως η δημόσια πίεση μπορεί να ε, αναγκάσει σε μετατόπιση σε τέτοιου ζητήματα. Ως προς το θέμα των αμερικανικών φόρων και των εταιριών που φεύγουν εκτός χώρας, στο εξωτερικό, αυτό ήταν πραγματικά ένα ψεγάδι του φορολογικού μα ε, συστήματο, το οποίο έπρεπε να έχει διορθωθεί. Το γνωρίζαμε από καιρό. Το γνωρίζαμε και λέγαμε ότι οι αμερικανικές ε, εταιρείες, οι αμερικανικοί όμιλοι που βγάζουν χρήματα, κερδίζουν χρήματα στο εξωτερικό, δεν φορολογούνται από το κέρδου εφόσον δεν το επαναφέρουν το κέρδος αυτό στι ΗΠΑ. Και αυτό βεβαίω είναι κίνητρο για να μην επενδύουν στι ΗΠΑ. Έπρεπε να βρεθεί ένα κίνητρο. Ήταν ε, ένα σύστημα που μα ε, έπλητε εσωτερικώ στο φορολογικό σύστημα. Και αυτό δείχνει το πόσο δυνατέ είναι και πολυεθνικέ βέβαια, έτσι. Ε, μπορούσαν αυτέ να πιέσουν ακριβώ και να περάσει στο φορολογικό μα σύστημα αυτό το στοιχείο ω ως μέτρο ε, για να δημιουργηθούν και θέσει απασχόληση ίσως τελικά. Πίεσαν επί αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ε, η ιστορία των φορολογικών σήμερα είναι ότι διακοπές έχουν. Διακοπές χωρίς το όφελος το οποίο αποσκοπούσαν. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής για το ΕΛΚ, ο κύριος Ντάριος Ροζάτη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στίγκλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας σήμερα. Η δική μου ερώτηση αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη έτσι ώστε να μειωθούν τα κίνητρα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες να πάνε σε φορολογικούς παραδείσους και να ε, δημιουργήσουν διάφορες εταιρείες ε, προπέτασμα, καταπιστεύματα, ιδρύματα κτλ. Τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε το φορολογικό μας σύστημα, να βελτιώσουμε τη φορολογική νομοθεσία για να μην υπάρχουν αυτά τα κίνητρα. Να μειώσουμε δηλαδή την έλξη που τους ε, ασκούν ε, αυτή η φορολογική παράδεση. Και άλλη μια ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα έτσι ώστε να ασκήσει πίεση σε ε, χώρες που δεν συμμορφώνονται έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα. Ε, χωρίς όμως αυτή η πίεση να θεωρηθεί πως παραβιάζει την εθνική τους κυριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, καθηγητά Στίγκλιτς, έχετε το λόγο. Η εθνική κυριαρχία είναι πάντα ε, κάτι το περίπλοκο. Πρέπει όμως να το συνδυάσουμε με την υπεύθυνη εθνική κυριαρχία. Όταν μια χώρα ε, κάνει πράγματα τα οποία βλάπτουν μια άλλη χώρα, αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι όταν ας πούμε μια κυρίαρχη χώρα μολύνει το περιβάλλον, συνεισφέρει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, τότε αυτό που κάνει είναι βλαβερό για τις άλλες χώρες. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο η φορολογική παράδειση βλάπτουν άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται να παραμείνουν ατιμόρυτες πράξεις οι οποίες είναι επιζήμιες για τη διεθνή κοινότητα, για τους πολίτες όλου του κόσμου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να μας ανησυχεί ε, αυτό που λέτε. Σίγουρα μία χώρα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί ας πούμε να ε, έχει και να θέτει πυρηνικά όπλα. Επίσης. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ασκήσουμε πίεση στα μη συνεργάσιμα κράτη έχω ένα μέτρο να προτείνω το οποίο μπορεί να θεωρείται ακραίο, όμως ε, ενδεχομένως να χρειαστεί να το λάβουμε. Για παράδειγμα, εάν μια χώρα δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα, να μην έχουν το δικαίωμα οι δικές μας εταιρείες των δικών μας ε, χωρών να δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή. Δηλαδή να μην, να μην ε, μπορούν οι δικές μας τράπεζες να συνεργάζονται με τις δικές τους. Είναι σαν ένα ιός φανταστείτε, σαν μια μολυσματική ασθένεια που προσπαθούμε να περιορίσουμε έτσι ώστε αυτή να μην εξαπλωθεί. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στις δικές μας τράπεζες να ε, συνδιαλέγονται, να συνεργάζονται με εκείνες τις τράπεζες των ε, κρατών που δεν συνεργάζονται. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Και αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε απάντηση. Αυτά τα εξωχώρια τραπεζικά κέντρα τι προσφέρουν στη διεθνή κοινότητα ως χρηματοπιστωτικά κέντρα. Ένας από τους υποψήφιους ε, προέδρους πριν από τέσσερα χρόνια μάλιστα είπε ανοιχτά ότι διατηρούσε λογαριασμού στις νήσους ε, Καϊμάν. Και μάλιστα αναφέρθηκε ε, το αν η Νέα Υόρκη είναι κατάλληλο τραπεζικό κέντρο και μάλιστα ότι επίσης η νήση Κέιμαν κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από το Λονδίνο, για παράδειγμα. Αλλά, ξέρετε, τα χρήματα δεν φυτρώνουν σε δέντρο το οποίο στις και Κέιμαν έχει περισσότερο ήλιο. Όχι. Το σκεπτικό, λοιπόν, πίσω από το να επιτρέπεται αυτό το φορολογικό και νομοθετικό αρμπιτράζ νομίζω πως πρέπει να αμφισβητηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σέτζιο Κομφεράτη έχει το λόγο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθηγητά, όπως τα γνωρίζετε μάλλον, έλεγα, όπως τα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να ετοιμάσει μια σειρά από νομοθετικά μέτρα ε, για τα φορολογικά. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω την ε, σημασία αυτών των προσπαθειών και των γραπτών σας απαντήσεων. Στις γραπτές σας απαντήσεις θίγεται το θέμα των λεγόμενων φορολογικών προτιμήσεων και των ζωνών που είναι αφορολόγητες και ότι θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτού του μηχανισμού. Συμφωνώ με το γεγονό ότι η απουσία φορολογία για τι εταιρείε ή, ή ο φόρο που είναι κοντά ή πλησιάζει στο 0, είναι 0, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα μαζί με το απόρριτο. Ώστε να δούμε τι θα γίνει με την ε, νομοθεσία ε, για τις περιπτώσεις των ε, εταιριών και προκειμένου να έχουμε τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Ευχαριστούμε. Ε, ναι. Είναι σημαντικό αυτό, το έλεγα και προηγουμένως, αλλά θέλω να επικεντρωθώ στο ρόλο των Εβραίων φορολογικών προτιμήσεων. ιδιαίτερως για αυτές τις φορολογητές περιοχές σε ορισμένε χώρες που επιτρέπουν πολλά κάποιες ασυμβοσίες Είναι μία ε, δυνατότητα για να υπάρχει λεύκανση παράνομων προσόδων, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Όταν περνάει κανεί σε χρηματοοικονομικέ δραστηριότητε, παριστάνει ότι κάτι κάνει, ότι παράγει κάποιο είδου ύφασμα λόγου χάρη, κάνει λίγο από αυτό και η βασική του δραστηριότητα είναι το ξέπλυμα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του να χρησιμοποιεί κανεί ε, τι αφορολόγητε περιοχέ είναι ότι το κέρδο δεν φορολογείται. Γι' αυτό υπάρχουν ε, τέτοιου είδου πρότυπα και προδιαγραφέ ακόμη και για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματο. Όπω ε, το στοίχημα, τα στοιχήματα και ο τζόγο. Αλλά όταν βλέπει κανεί ε, δραστηριότητε ξεπλήματο σε αφορολόγητε περιοχέ πρέπει να τι εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε που είναι νομότυπε ή νόμιμε, αλλά μπορεί να υπάρχει και πραγματικό ξέπλυμα. Γι' αυτό λέω ότι τα πρότυπα όσων λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές και έχουν δραστηριότητες θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτά όλα αυτά σε όποιον θέλει να αναλάβει δραστηριότητες εκεί. Σε αυτές τις περιοχές όποιος έχει οποιαδήποτε αξιόμενη δραστηριότητα θα πρέπει να μην επιτρέπεται να δραστηριοποιηθεί. Και αν το επιτρέπει η κυβέρνησή του, θα πρέπει να μπαίνει κατευθείαν σε μαύρη λίστα. Δεν παίρνει κανεί άδεια να ανοίξει τράπεζα αν είναι ένα χαρακτήρα ε, που δεν είναι διπόληπτο. Αυτό είναι προδιαγραφή σε κάθε χώρα για να πάρει κανεί άδεια να βρει μια τράπεζα. Δεν μπορεί κανεί με κακό ιστορικό να ανοίξει τράπεζα όλες οι δραστηριότητες αναγκαστικά θα βασιστούν σε αυτήν την άδεια για την ε, ίδρυση τράπεζας και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για όσους ε, λειτουργούν σε αφορολόγητες περιοχές. Thank you Ευχαριστώ πολύ ο επόμενος ομιλητής. Είναι ο καθηγητής Μπέρντ Λούκε από το CCCR. Καθηγητά Στίκλιτσεν, κατάλαβα σωστά αυτό που μας συστήνεται είναι να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Επί αυτό ακριβώ εργαζόμαστε εδώ. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το νομικό τοπίο έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια. Τώρα είστε οικονομολόγος, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω για δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή για τις επιχορηγήσεις και τα κίνητρα. Και τα αρνητικά κίνητρα. Το σύστημα όπως λειτουργεί το σύστημα, από ό,τι το κατανοώ, είναι πως έχουμε μια λυσίδα ανθρωπών που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Υπάρχουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, υπάρχουν οι χρηματοπιστωτικοί σύμβουλοι στις τράπεζες και στους χρηματοπιστωτικού θεσμούς. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νομικές εταιρείες στον Παναμά και αλλού στον κόσμο και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι όντω λειτουργούν τις υπερακτίες εταιρείε. Η ερώτησή μου είναι πως εάν αυξήσουμε τη διαφάνεια και σπάσουμε τη γραμμή αυτή των ανθρώπων σε ένα σημείο, τι πιστεύετε για δυνατότητες υποκατάστασης, για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Με ποιους τρόπους θα βρουν νέους μηχανισμούς για να αποκρύψουν τα φορολογητέα τους έσοδα, υποκαθιστώντας παραδείγματος χάρη τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες. Η δεύτερη ερώτηση είναι, τι πιστεύετε για την μείωση των κινήτρων φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής ή για την αύξηση κινήτρων στους πληροφοριοδότες, ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα φαινόμενα αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Έτσι οι εταιρείε δεν θα μπορούν απλά να αποχωρούν με την ευημερία που έχουν αποκτήσει. Αυτές οι δύο ερωτήσεις μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Πιστεύω πως έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια τεράστια εφοδιαστική αλυσίδα υπό την έννοια της παραγωγής αυτής της μυστικότητας σε αυτού του απορρίτου. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πως πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό σε όλα του τα σημεία. Εμεί προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε στο τουαρβιστικό σύστημα και εκεί προοδεύουμε. Αλλά διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν αρκεί. Γι' αυτό και τώρα προσπαθούμε να επιτεθούμε στο σύστημα αυτό, στο επίπεδο των νομικών εταιριών, των πραγματικών ιδιοκτητών και την αποκάλυψή τους. Και ελπίζω πως θα το αντιμετωπίσουμε και θα το καταπολεμήσουμε σε αρκετά σημεία, σε αρκετούς κρίκους της αλυσίδας, έτσι ώστε να πετύχουμε τη διαφάνεια. Οι δυνάμεις υπέρ της μυστικότητας είναι αρκετά δυνατές ώστε να βρουν κάποιον άλλον τόπο. Γι' αυτό και τονίζω πως, πως πρέπει να είναι μια παγκόσμια επίθεση κατά του συστήματος αυτού. Για μένα δεν είναι προφανές πως αν επιτεθούμε με τον τρόπο που ανέφερα, όντως θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό. Πιστεύω όμως πως οι χειρότερες πτυχές που αποκαλύφθηκαν από τα Panama Papers, αυτές τουλάχιστον μπορούμε να τις εξαλείψουμε. Είμαι αισιόδοξο ως προς αυτό. Και αν δεν τα καταφέρουμε, αν έχουμε έρευνες από αυτή την επιτροπή ή από άλλες, τότε θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε και τις νέες μορφές που θα λάβει το φαινόμενο αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουν μυστικότητα σχετικά με τη μυστικότητά τους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν και αν προσπαθήσουμε πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε. Το δεύτερο, στο οποίο συμφωνώ και πάλι, ναι, χρειαζόμαστε κίνητρα για πληροφοριοδότες. Πιστεύω πως αυτό βοηθάει. Αυτό που με ανησυχεί και το οποίο περιέχει και η έκθεση είναι πως σε κάποιες χώρες Συμβαίνει το αντίθετο. Πληροφοριοδότες μπορεί να φυλακιστούν. Και μια χώρα με ένα νομικό πλαίσιο όπως αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στη μαύρη λίστα. Δηλαδή κάποια από τα πράγματα τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν στη μαύρη λίστα είναι νομικά πλαίσια τα οποία δυσχεραίνουν τη διαφάνεια. Αυτά με τέτοια αρνητικά κίνητρα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όπως αυτή η νομοθεσία που ποινικοποιεί τους πληροφοριοδότες. Πρέπει να διασφαλίσουμε οι χώρες να μην έχουν τέτοιους νόμους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάιτε Ρουίς από την Άλτε. Ε, muchísimas gracias, σας ευχαριστώ πολύ, καθηγητά Στίγκλιτς. Αυτό το κοινοβούλιο έχει μια ιστορική ευκαιρία για να πατάξει αυτά τα φαινόμενα. Είναι φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, διαφθορά. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση. Χρειαζόμαστε κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει υποβάλει μια πρόταση για μια τέτοια μαύρη λίστα στην Ευρώπη. Και πιστεύω πως ε, το θέμα της εταιρικής παφορολογίας θα μπορούσε να ε, συζητηθεί έτσι ώστε να συνεισφέρει σημαντικά σε μια αλλαγή. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ε, κριτήριο. Εσείς θεωρείτε πως αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση. Και μια άλλη ερώτηση. Τι θεωρείτε ποια είναι η άποψή σας για τα επόμενα, ε, τα υπόλοιπα κριτήρια που θα ε, ισχύουν για να μπει κάποια εταιρεία σε αυτή τη μαύρη λίστα. Η Γερμανία και το Λουξεμβούργο βρίσκονται αρκετά ψηλά σε αυτήν την λίστα ε, φόρο αποφυγής. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι θα επιθυμούσαμε να σας βλέπουμε πιο συχνά γιατί σίγουρα θα βοηθήσετε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθηγήτα Στίγκλιτς, έχετε το λόγο. Όπως είπα και πριν, εδώ είναι πολλοί παράγοντες. Πιστεύω πως ο μηδενικός εταιρικός φόρος είναι κάτι το οποίο είναι συνυπεύθυνο για αυτό το φαινόμενο, για αυτόν τον ανταγωνισμό που οδηγεί στην φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Η Διεθνής Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση του, της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας, της οποίας πρόεδρος είναι ο Αντώνιο, έχει δημοσιεύσει μία μελέτη η οποία εστιάζει στη, στον ανταγωνισμό τον φορολογικό. Και εάν επιτρέψουμε αυτό το φαινόμενο να συνεχίσει να εξαπλώνεται, τότε οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Η μηδενική φορολογία για τις εταιρείες, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να βρεθούν κάπου αλλού και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να επομιστούν αυτό το φορτίο. Δυσανάλογα. Τώρα, το θέμα της μηδενικής φορολογίας σε συνδυασμό με το φορολογικό απόρριτο και το ξέπλυμα χρήματος, ε, σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπα και πριν. Όμως, δεν, δραστη... δεν ε, συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες όλες οι χώρες που έχουν μηδενική φορολογία. Δεν συμμετέχουν σε αυτόν τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό. Όμως, όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι μηδέν, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι σημαίνει αυτό. Όταν δεν έχεις έσοδα, αφού η φορολογία είναι μηδενική, πού θα βρεις τα λεφτά. Πολλές φορές οι επιπτώσεις είναι στις θέσεις απασχόλησης. Και όπως στην περίπτωση της Apple, με την Ιρλανδία, δημιουργήθηκαν ελάχιστες θέσεις εργασίας από την Apple στην Ιρλανδία, ακριβώς ε, επειδή υπήρχε αυτή η μηδενική φορολογία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναρτηθούμε ε, τι γίνεται. Τι θα μπορούσε τώρα να κάνει η Ευρώπη εντός των συνόρων της. Θα μπορούσε όλες αυτές οι φορολογικές συμφωνίες να δημοσιοποιηθούν. Γιατί δηλαδή η Apple να έχει διαφορετική μεταχείριση από την General Electric, ας πούμε, από την Google, από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Αυτό συνέβη μόνο εξαιτία ε, του Αμερικανικού Κογκρέσου, το οποίο ανακάλυψε ότι η Apple είχε μία ειδική συμφωνία. Και αυτή η μυστικότητα έχει ως επακόλουθο το να μην υπάρχει πληροφόρηση. Και όπως σας είπα, εξαιτίας του Αμερικανικού Κογκρέσου μάθαμε όλοι τι γίνεται στην Ιρλανδία. Αυτό δεν πρέπει να είναι ανεκτό. Όλες οι συμφωνίες πρέπει να είναι δημόσιες, έτσι ώστε να έχουν όλη πρόσβαση και να μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενό τους και να δουν εάν υπάρχει κάποια ειδική συμφωνία, είτε για την Apple, είτε για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι εάν οι συμφωνίες αυτές ήταν δημόσιες, τότε θα ζητούσαν και άλλες εταιρείες ειδική μεταχείριση. Και αν και άλλες εταιρείες ζητούσαν ειδική μεταχείριση, τότε τα φορολογικά έσοδα της Ευρώπης θα ήταν μηδέν. Μηδέν από όλες τις αμερικανικές εταιρείες. Στη συνέχεια, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα δεχόταν τη συνέχεια αυτών των συμφωνιών Γι' αυτό λοιπόν όπω καταλαβαίνετε υπάρχουν βαθύτατες πολιτικέ συνέπειε σε αυτές τις πρακτικές και είμαι βαθύτατα απογοητευμένο από το ότι μία χώρα, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί με τέτοιο τρόπο τι υπόλοιπε. Σα ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Φάμπιο Τιμάζη από την ΚΟΕ. Καλώ ήρθατε κυρίε Στίγκλιτ. Μόλι αναφέρατε την Ιρλανδία και η Ιρλανδία ανέφερε 26% ανάπτυξη πρόσφατα χάρη στο φορολογικό τη μοντέλο. Το πρόβλημα όμω είναι ότι ο μέσο Ιρλανδό πολίτη δεν είδε κάτι από αυτό. Μπορείτε να εξηγήσετε συνεπώ, πώ πιστεύετε πω θα συμβάλλει η φορολογική δικαιοσύνη στην στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της Ευρώπης, όπως είναι η έλλειψη ανάπτυξης και η λιτότητα. Μπορεί να παίξει θετικό ρόλο για την οικονομική ευημερία των πολιτών μας. Δεύτερον, όταν μιλούμε για μια μαύρη λίστα, όταν πήγαμε στην Ουάσιγκτον με την προηγούμενη Επιτροπή μας υπόθηκε πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τον Delaware ή άλλες πολιτείες επειδή μπορούμε να ασχοληθούμε με φορολογικούς συντελεστές αλλά όχι με την ομοθεσία περί απορρίτου. Πιστεύετε πως μπορεί να πιστεί ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι σχετικά με αυτό. Δηλαδή να μπει το Delaware στην λίστα των στη λίστα των φορολογικών παραδείσων. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω από τη δεύτερη ερώτηση. Ναι, θα βοηθούσε πολύ να επιβάλλεται κυρώσεις ενάντια στο Delaware ή όπου αλλού υπάρχουν πολιτείες στην Ευρω... στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν συμμορφώνονται. Μου φαίνεται λοιπόν πως μπορεί να υποθεί πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο δικαιοδοσίες που υιοθετούν συγκεκριμένα πρότυπα. Οι συγκεκριμένες δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά και μπορείτε να πείτε πως λυπούμαστε. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν μπορούν να συνεργαστούν με τράπεζες ή με πολιτείες των ΗΠΑ που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά. Αυτό σίγουρα και θα επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα και πιστεύω πως θα αλλάξει τη συμπεριφορά τους. Πιστεύω πως αυτό που ακούσατε από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν παρά μια δικαιολογία το ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Για παράδειγμα λοιπόν, αυτό έρχεται εν μέρει ως απάντηση στην οργή που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν περιπτώσεις ε, αγορε, αγορών διαμερισμάτων αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου από εταιρείε τους ιδιοκτήτες των οποίων δεν γνωρίζαμε. Ήταν ξεκάθαρο λοιπόν, πολύ ξεκάθαρο, πως εκεί τουλάχιστον υπήρχε η υποψία ξεπλήματος χρημάτων σε μαζικό βαθμό στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η κυβέρνηση αντέδρασε δηλώνοντας ότι θα πρέπει να αποκαλυφθεί η πραγματική κυριότητα των εταιριών αυτών στο City της Νέας Υόρκης αλλά και στη Ουάσιγκτον. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αν ήθελε. Γι' αυτό και πιστεύω πως οι κυρώσεις θα συνέβαλαν, θα, θα ενθάρρυναν την κυβέρνηση να λάβει πιο δραστικά μέτρα και θα βοηθούσαν πολύ. Το ευρύτερο ζήτημα που θέσατε, πρώτα απ' όλα, όταν μιλάτε για 26% ανάπτυξη στην ε, Ιρλανδία, πιστεύω πως όλοι γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι πραγματικό. Δεν υπάρχουν χώρες που σημειώνουν ανάπτυξη της τάξης του 26%. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό για αυτό που συμβαίνει. Μπορεί να έχουμε αύξηση 26% του δηλωνόμενου ΑΕΠ αλλά οι πολίτες της Ιρλανδίας φυσικά και δεν πλούτησαν κατά 26%. Σίγουρα θα υπάρχουν και στοιχεία για τους ανθρώπους. Ε, και αν ψάξετε να βρείτε κάποιον τα εισοδήματα του οποίου αυξήθηκαν κατά 26% το περασμένο έτος, σίγουρα δεν θα βρείτε σχεδόν κανέναν. Και αυτό δείχνει στην κλίμακα των δραστηριοτήτων φόρο αποφυγής. και της οικονομικής δραστηριότητας. Αλλά το γενικότερο θέμα που θέσατε είναι πως όταν δεν υπάρχουν πραγματικά φορολογικά έσοδα, λόγω όλων αυτών των περίεργων συναλλαγών, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κόστος επειδή δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές, στην παιδεία, στην τεχνολογία που χρειάζονται για την πραγματική ανάπτυξη, όχι για την εικονική όπως την είδαμε στην Ιρλανδία, αλλά για την πραγματική που αυξάνει την, τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Αυτό δεν γίνεται χωρίς επενδύσεις. Γι' αυτό και το ζήτημα εδώ είναι η προοπτική της Ευρώπης αλλά και του κόσμου στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ καθηγητά Στίκλιτς. Για τους πρασίνους, ο Πασκάλ Ντυρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, καθηγητά Στίκλιτς. Είστε ένας οικονομολόγος παγκόσμιας φήμης. Είσαστε και γνωστός κονσάλταντ, αλλά όχι μόνον. Είσαστε και ένα προεξέχον ε, μέλος, ένα γνωστό μάλλον ε, μέλος της κυβέρνησης Κλίντον επί τέσσερα χρόνια. Βέβαια, οι ψηφοφόροι αποφάσισαν διαφορετικά. Ε, αλλάζουν οι καιροί και ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις οι οποίες είναι κάπως αλληλένδετες με την προσωπική σας πορεία. Η πρώτη είναι αυτό που είπατε πολύ ξεκάθαρα. Χρειάζονται κυρώσεις. Χρειάζεται όσοι δεν σέβονται τους κανόνες να ε, τιμωρούνται. Ε, εδώ θέλω τη γνώμη σας για την ήπια ρύθμιση την υπερνοθεσία και την αυτορύθμιση. Διότι τα δικαιωτικά γραφεία, οι εισαγγελεί έχουν κανόνε. Εσεί για ποιου κανόνε μιλάτε, ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι, ε, τι είδου περιορισμού θα επιβάλλουμε, πώ θα εφαρμόζονται αυτά, επειδή έτσι κι αλλιώ διατάξει και μέτρα υπάρχουν. Και δεύτερη ερώτηση, πολύ σύντομα. Βρεθήκατε πολύ κοντά και ακριβώ στην καρδιά των ενδιαφερόντων των ε, ηθινόντων. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, γιατί τα προβλήματα τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη που υπάρχουν εδώ και χρόνια, γιατί εμποδίστηκαν οι ηθήνοντες να εφαρμόσουν δημόσιες πολιτικές, κρατικές πολιτικές, οι οποίες θα βάλουν τέρμα σε αυτές τις πρακτικές. Ευχαριστούμε καθηγητά Στίγκλιτς. Σε πολλούς τομείς η ήπια νομοθεσία μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο. ε, ανέπτυξε το επιχείρημα ότι για την εξυγίανση του κρατικού χρέους λόγω χάρη θα είναι ένα πολύ καλός τρόπος. Ε, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει με την κλασική νομοθετική διαδικασία. Θα είναι πολύ αυστηρός ο τρόπος αυτός. Ήδη σε πολλούς κλάδους υπάρχει υπερνομοθεσία, πολλές ε, πιέσεις, αλλά δυστυχώς στη φοροδιαφυγή φάνηκε ότι είναι ανθεκτικό το φαινόμενο. Επιβιώνει ό,τι και αν λέει ο κόσμος η ανοιχτή παρουσίαση, η διαφάνεια ε, δεν καταργεί αυτά τα, αυτούς τους λιμένες απορρίτου. Δεν τους αρκεί η πίεση της ήπιας νομοθεσίας. Γι' αυτό κάποιος πρέπει κανείς να αυξήσει την ένταση, την άσκηση πίεσης. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ως προς την προ τα θέματα για τα οποία μιλάμε. Για πολλά από αυτά υπάρχουν πρότυπα, υπάρχουν διατάξει και νόμοι που οι δικηγόροι τα γνωρίζουν. Θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι καινούριο, όντω. Απλώ πρέπει να υλοποιήσουμε τα πρότυπα που ήδη έχουμε. Για παράδειγμα, συνεργός σε παιδική πορνεία. Αποδείχτηκε συνέργεια και σε αυτή την περίπτωση με το Panama Papers. Ξέρουμε ότι το να είναι κανείς υποκινητής και ε, να επιτρέπει, να υποθάλπει τέτοιου είδους δραστηριότητε είναι παράνομο. Οποιοςδήποτε είναι παράνομος. Οπότε κάποια στιγμή αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να επιβάλλουμε νόμους και πρότυπα που ήδη έχουμε. Όμως προφανώς δεν το κάνουμε. θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτούς τους ε, λιμένες απορρίτου. Καταλαβαίνοντας ότι ακόμα και αυστηρή νομοθεσία να υιοθετήσουμε, την κλασική δηλαδή, όχι καν την ήπια, ούτε καν μάλλον την ήπια, ήδη θα είναι δύσκολο να αποτύχουμε αποτέλεσμα. Οπότε πραγματικά χρειάζεται σοβαρότερη επιβολή και ίσως και υψηλότερα πρότυπα διότι πάντοτε θα προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Και βελτιώνοντας τα πρότυπα μπορεί να είναι σαφές πια ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια που έχουμε θέσει με τις συμπεριφορές τους. Οπότε εκεί ίσως να εντοπίζονται. Για τα εμπόδια που ρωτήσατε και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι λύσεις θα μπορούσαμε να βρούμε γι' αυτά. Θα έλεγα είναι δυο λογιών. Πρώτα απ' όλα η αδράνεια και το άλλο οι ομάδες πίεσης. Παράδειγμα για την κάθε περίπτωση. Όταν ήμουν στην κυβέρνηση Κλίντον, έθεσα το ζήτημα του συστήματος μεταφοράς τιμών Ένα σύστημα διεθνούς φορολογίας για τις πολυεθνικές θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει. Η αντίδραση των ε, ανθρώπων του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι έχουμε προσπαθήσει πολύ ε, σκληρά για να έχουμε ε, αυτό το σύστημα με τα παραστημόνα από το 1920. Δεν θέλουμε να αλλάξει. Ήδη μας είχε εξαντλήσει τη δεκαετία του 20 η προσπάθεια αυτή. Αυτό ονομάζω αδράνεια ακινησία. Δεν ήθελαν να αλλάξει τίποτα στις ζωές τους. Και δεν το θεωρούσαν καν σημαντικό. Εγώ το θεωρούσα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν μπορούσα να τους ε, βάλω συρτούς να το κάνουν. Τώρα καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα πλέον. 25 χρόνια μετά το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί. Ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε τότε, ε, δεν λειτουργεί και τώρα. Η ένταση λοιπόν έχει αυξηθεί και ελπίζουμε ότι με τη Διεθνή Επιτροπή που έχει αναφέρει και ο Χωσέ Αντώνιο στην οποία συμμετέχει ο Χωσέ Αντώνιο, θα υπάρξει καλύτερο φωτισμό του όλου θέματο. Αυτό ήταν η αδράνεια. Και έπειτα προφανώ οι ομάδε άσκηση πίεση. Για του περισσότερου από αυτού του τομεί, κάποιοι προφανώ υποφελούνται από τι τωρινέ διευθετήσει. Και όσοι υποφελούνται δεν θέλουν να χάσουν τα ωφέλη του. Τόσα απλά τα πράγματα. Άλλο ένα παράδειγμα. Τελείω διαφορετικού χαρακτήρα. Προσπάθησα να περάσω ένα μέσο πράσινου ΑΕΠ για να αποφύγουμε την υποβάθμιση των μέσων και την ε, καταστροφή των πόρων. Ξέρω ότι ήταν σημαντικό, αλλά η βιομηχανία του άνθρακα, το λόμπι του Άρθρακα στο Κογκρέσο, είπε ότι άμα συνεχίσω να λέω τέτοια θα μας πάρουν όλο το χρήμα. Μάλλον κάπου χτύπησα στα νεύρα κάποιου, πάτησα κάποιο κάλο και προφανώς δεν ήθελαν να επικεντρωθεί η προσοχή της κοινή γνώμης στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω του άνθρακα. Πολλοί βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή την ε, ιστορία και από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη με τις τωρινές διαθετήσεις προφανώς κερδίζουν. Εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Ευχαριστούμε. Πρέπει να κοιτάμε και το ρολόι, διότι έχουμε μόνο 7 λεπτά αλλά πολλούς ομιλητές. Θα πρέπει να συντομεύσουμε και στις ερωταπαντήσεις και στις απαντήσεις παρακαλώ. Επόμενος ομιλητής, ο Ray Finch από τους EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθηγητά Στίγκλιτς, στην έκθεσή σας για την ε, παραοικονομία και για κάποια στοιχεία των φορολογικών παραδείσων λέτε ότι το απόρριτο θα πρέπει να έρθει από το διεθνές, φορο... από το διεθνές χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα. Και λέτε εκτός και αν πληρώνουν οι εξής προποθέσει. Δηλαδή, στο τρίτο σημείο αναφέρεται ότι πρέπει κάθε τράπεζα να αποκαλύπτει την αλληλογραφία ή τι επαφέ που έχει με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή κάποια, α, κάποιον όμιλο που μπορεί να μην είναι εταιρεία. Τι εννοείται ότι θα πρέπει η αμερικανική νομοθεσία να διαφέρει από τον υπόλοιπο κόσμο, ε, ότι θα πρέπει να Ε, συμμορφούνται όλοι με αυτές τις προδιαγραφές και να τιμωρούνται οι κανονικοί άνθρωποι. Και επίσης, πώς θα σχολιάζεται όσα είπε η κυρία Κλίντον για τις σχέσεις με πολυεθνικές στη Μέση Ανατολή που μπορεί να χρηματοδότησαν την πολιτική της σταδιοδρομία και εκστρατεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για το ζήτημα των χωρών που κερδίζουν, υπονομεύοντας το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχω την εντύπωση ότι το απέντησα προηγουμένως, ε, απαντώντας τον κύριο Ροζάτη για την ε, εθνική κυριαρχία. Υπάρχει ένα θέμα υπεύθυνη, υπάρχει μια μια διάσταση υπεύθυνη κυριαρχία και μια άλλη που επιβάλλεται ει βάρο άλλων. Αυτή η χώρα θα πρέπει να είναι πρόθυμη να πληρώσει και το κόστο, το τίμημα. Και θα πρέπει οι πολίτε αυτή τη χώρα να λένε ότι. να λένε στην κυβέρνησή του δεν μπορείτε να, επιβάλλετε, να επιβάλλετε το κόστος σε άλλους, δεν μπορείτε να γλιτώνεται με, να τις καπουλάρετε με την ε, ρήπανση, με τις κλιματικές αλλαγές, με περιπτώσεις όπως η παιδική πορνογραφία, οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες έχουν κόστος. Έχουν κόστος που επιβάλλουμε στις υπόλοιπες κοινωνίες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς, όταν επιβάλλεται κόστος σε άλλες χώρες, ε, θα υπάρξουν και θύματα. Αυτό είναι η συνέπεια οποιασδήποτε μορφής, οποιασδήποτε μορφής κυρώσεων. Επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία. Ε, είδατε τι έκανε η Ρωσία. Κατέλαβε την Ανατολική Ουκρανία. Ο ομιλητής. Ο κύριος Λεμπρετών από την ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ κύριε Στίγκλιτς ε, στην ευχαριστώ που ήρθατε στην Εξεταστική Επιτροπή. Ε, το ερωτηματολόγιο από την Επιτροπή μας έδειξε ότι τρίων ειδών ε, οικονομικά εγκλήματα διαπράχθηκαν. Πρώτα απ' όλα αυτά που αφορούν εταιρείε. Δεύτερον, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από, από το οργανωμένο έγκλημα. Και δεύτερον, η απόκρυψη ε, του οικονομικού εγκλήματος ε, υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης από πολλά κράτη. Και την τρίτη περίπτωση. Θεωρείται ότι ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολεμούν δραστικά με τη διαφθορά, διαθέτουν τα εργαλεία για να το κάνουν αυτό, αλλά δεν το πράττουν. Έχω λοιπόν τι εξή ερωτήσει. Πρώτον, πιστεύετε ότι η εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ θα φέρει τι ΗΠΑ στην ανάγκη να, να κάνουν εντονότερε μεταρρυθμίσει. Δεύτερον, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να καταπολεμήσει την προδιαφυγή και τη φοραπάτη, ενώ ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει πρόεδρο ενό φορολογικού παραδείσου, ε, τον, ε, του Λουξεμβούργου τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Και τρίτον, δεν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη περισσότερο ε, με το ευρώ από ό,τι αν υπήρχαν τα εθνικά νομίσματα. Τέσσερα, η διαφθορά και η φοροαπάτη δεν είναι αποτέλεσμα της, ε, του διεθνού ε, νεοφιλελευθερισμού. Μήπω πρέπει να επανέλθουμε σε έναν οικονομικό συντηρητισμό για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Ευχαριστούμε για αυτήν την δήλωση. Η δεύτερη ερώτηση έχει ήδη απαντηθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που θίξατε το τρίτο σημείο, το απόρριτο. Έχει να κάνει και με τους συγκρισίους συμφερόντων και την διαφθορά και στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις προηγμένες οικονομίες. Είναι μια μεγάλη πηγή προβλημάτων. Όταν ήμουν ένα από του βασικού οικονομολόγου τη Παγκόσμια Τράπεζα, ήταν από του προβληματισμού μου αυτό. Ε, μαζική διαφθορά σε πολλέ χώρε υπήρχε και πολλοί από το χρήμα το κρύβαν στο Λονδίνο. Εκεί δεν μπορούσαν να το πάρουν πίσω αυτέ οι χώρε που θέλανε. Αυτό είναι ο ρόλο του Λονδίνου. Έτσι λειτουργεί ο λιμένα απορρίτου. Ανησυχώ ιδιαίτερω λοιπόν, ανησυχώ με την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ ανησυχώ διότι όλα αυτά θα γίνουν λίγο πιο αδύναμα, θα υπάρχει λιγότερη δίωξη, πιο αδύναμη δίωξη. Και το απόρριτο μπορεί να παραμένει. Δεν έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Όμως, όπως ε, σωστά εντοπίσατε, Γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως ηγέτη αρχιτέκτονα του συστήματος φοροδιαφυγής και φοραπάτης και αυτό προφανώς έχει πλήξει και έχει ζημιώσει άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά το γνωρίζει τόσο καλά ο κόσμος που ευτυχώς έχει προκαλέσει προσοχή, την προσοχή και το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Και το γεγονός ότι το ερώτημα τίθεται θα πει ότι βρίσκεται παρόν στο νου της κοινή γνώμης. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα που δεν μπόρεσα να θίξω και τα οποία θα διευκόλυναν και διευκολύνουν την διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας. Το ένα είναι ότι ο είναι οι μετοχές του κομιστή, λεγόμενες μπέρεσες. Και επίσης με τα χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας. Μειώνεται το κόστος του να κουβαλάει κανείς χρήματα πάνω του. Ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος, αλλά πρέπει να πω μια σύντομη ιστορία. Δηλαδή, όταν ε, ήμουν στο Συμβούλιο των ε, Οικονομολόγων, Ήθελα να γλιτώσουμε τα αμερικανικά ομόλογα στον κομιστή, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παρόμοιους σκοπούς, για διαφθορά. Και η απάντηση των ανθρώπων του Υπουργείου Οικονομικών μου λέγανε άμα τα καταργήσουμε θα αυξηθούν τα επιτόκια. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι λένε ότι η ζήτηση αμερικανικών ομολόγων είναι από αυτούς που θέλουν αδιαφάνεια και να αποφύγουν τους φόρους και είναι τόσο μεγάλη που επηρεάζουν τι τιμέ. Χάνει κανεί όμω φορολογικό εισόδημα δίνοντα τα ομόλογα. Δηλαδή από τη μια κερδίζει από την άλλη χάνει. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο συνένοχοι σε αυτή τη διαφορά. Κι όμω το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επικεντρωνόταν λαθασμένα στο θέμα του να ελεγχιστοποιήσω τα επιτόκια. Μάλλον προκειμένου να μην ελεγχιστοποιηθούν τα επιτόκια να δεχτούμε τη διαφθορά και τη φοροαποφυγή. Για μένα ήταν πραγματικά ένα συλλογισμό που δεν μπορούσα να καταπιώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ο προστατευτισμό είναι η απάντηση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πάει τα πράγματα πουθενά. Ήδη βρισκόμαστε σε ένα κόσμο αρκετά ενοποιημένο, ο κόσμος κυκλοφορεί αρκετά και ο προστατευτισμός δεν είναι απάντηση. Η ορθή απάντηση είναι όταν έχουμε εμπορικέ συμφωνίε να βεβαιωνόμαστε ότι οι εμπορικέ συμφωνίε συμπεριλαμβάνουν διατάξει που την διαφάνεια την ε, ε, βάζουν μπροστά. Και θα πρέπει να είναι ένα απόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε εμπορική συμφωνία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε δύο πρόσθετες ερωτήσεις από τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες, Γιούριτ Νίτερ Μάιερ και Εμμανουέλ Μορέλ. Λούντεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καθηγητά Στέγκλιτς που ήρθατε εδώ. Η πρώτη μου ερώτηση σχετίζεται με τις απαντήσεις σας σε ερωτήσεις της Επιτροπής. Μου φαίνεται πως όταν περιγράφεται τα δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν στον Παναμά και όχι μόνο εκεί, πως οι νομικές εταιρείες είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία επειδή οι τράπεζες και οι σύμβουλοι υπόκεινται σε, σε κάποιες ρυθμίσεις ενώ οι νομικές εταιρείες όχι. Αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι σωστή η παρατήρηση αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι η Επιτροπή αυτή εστιάζει στην φοροαποφυγή αντί για την φοροδιαφυγή. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε εσείς ότι ο οικονομολόγος πως το πολύ πολύπλοκο σύστημα των φορολογικών νομοθεσιών παίζει κάποιον ρόλο στα φαινόμενα αυτά για τα πόσο θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερο, περισσότερες προσπάθειες για την αποσαφήνιση των νομικών κειμένων. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά Στίγλιτς. Ναι, πιστεύω πως ένα από τα πιο από τους πιο αδύναμους της αλυσίδας σήμερα είναι οι νομικές εταιρείες. αλλά επίσης οι επιχειρήσεις, τα καταπιστεύματα, τα ιδρύματα με το απόρριτό τους. Εκεί πρέπει να μάθουμε την πραγματική κυριότητα. Αυτά πιστεύω είναι τα δύο αδύναμα σημεία του σημερινού πλαισίου. Συμφωνώ, η φόρο αποφυγή είναι μεγάλο πρόβλημα. μια πλούστευση θα ήταν μια προσέγγιση. Αλλά πάντα πρέπει να σταθμίζουμε, επειδή μπορούμε να απλοποιήσουμε τους φορολογικούς μας κώδικες, αλλά με μηδενική φορολογία θα έχουμε και μηδενική φοροδιαφυγή. Αυτό ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα της δημιουργίας φορολογικών εισόδων. Γι' αυτό και πρέπει να σταθμίζουμε πως αφενός επιχειρήσεις δείχνουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό ευφυΐας, εξυπτάδας. Με ένα πολύ έξυπνο φορολογικό σύστημα μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα βρουν έναν τρόπο να το κάνουν πιο πολύπλοκο και τον τρόπο αυτό δεν θα μπορείτε να το σκεφτείτε εκ των προτέρων. Υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας φορολογικών δικηγόρων εκεί έξω. Και όλοι, ένα μεγάλο μέρος της πολυπλοκότητας που υπάρχει, υπάρχει επειδή κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν τρόπους για να μην πληρώνουν φόρους. Ίσως υπάρχουν τρόποι. Περαιτέρω απλούστευσης μέσω επανεκκίνησης. Εάν αντιληφθούμε πως ο, ο δρόμος που έχει πάρει το σύστημα έχει αλλάξει πορεία λόγω παρεμβάσεων. Έχει αλλάξει πολλές φορές πορεία λόγω διαδοχικών παρεμβάσεων. Ίσως σε κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Ίσως πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εδώ και να ξαναγράψουμε τους κανόνες και να ξαναρχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής, Εμμανουέλ Μορέλ, 12 36. όπως διαπιστώσαμε όταν εξετάσαμε τις σχέσεις μας με τον Παναμά και όχι με τον Παναμά, πως το ξέπλυμα χρήματος και η φορολογική απάτη γίνονται μέσω εμπορικών συνδιαλλαγών. Τι πιστεύετε, πρέπει να υπάρχουν φορολογικές προϋποθέσεις σε σύμφωνα εμπορίου, εάν δεν έχουμε κάποιο κεντρικό μητρό των ιδιοκτητών εάν δεν το κάνουμε, τουλάχιστον αυτοί να μην επωφελούνται από τα σύμφωνα εμπορίου. Αυτό θα ήταν δυνατόν. Και δεύτερον, ναι, διάβασα τα κείμενα για το ευρώ. Ό,τι άποψη και να έχουμε για το ευρώ, για την περίπτωση της νομισματικής ένωσης χρειάζονται κάποια δίκτυα ασφαλείας για την φορολογική ασφάλεια. Σίγουρα αναζητάμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τη φοροαπάτη. Όμως, εάν υπήρχε ένας πραγματικός ελάχιστος συντελεστής ε, για όλες τις εταιρείε ε, στην Ευρωζώνη, δεν θα ήταν ένα σκόπιμο μέτρο για να μπορέσουμε να, να χαιρετήσουμε κάπω αυτή την ε, φοροδιαφυγή. Δυστυχώ δεν μπορούμε να συζητήσουμε την ε, κατάσταση του ευρώ σήμερα. Παρακαλώ. Συμφωνώ. Οι όρες της εμπορικές συμφωνίες είναι λόγοι για να ικανοποιηθούν οι βασικοί όροι αυτών των ευνοϊκών διευθυντήσεων. Αυτή είναι η αρχή της διαφάνειας. Επίσης, Βλέπετε στην έκθεση αυτή τέσσερις τρόποι για να αντιμετωπιστεί ο φορολογικός ανταγωνισμός. Πρώτη σύσταση της Επιτροπής μας είναι φορολογικός ανταγωνισμός να συμφωνήσουμε έναν ελάχιστο συντελεστή όντω για τις εταιρείε. Και περιγράφουμε πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο. Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούσαν σε ένα ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, αυτό τουλάχιστον θα δημιουργούσε ένα δάπεδο φορολογία. Ένα κατώτατο όριο. Και τέλο πάντων οι ακρότητε φοροδιαφυγή και φραπάτε που βλέπουμε δεν θα υπήρχαν. Ευχαριστούμε πολύ, καθηγητά Στίγκλιτ. Είναι προφανέ ότι η πείρα σας την οποία μοιραστήκατε μαζί μα σήμερα, είναι συναρπαστικού περιεχομένου για τη δουλειά της Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τρομερά πλούσια η συζήτησή μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνεί που εργάστηκαν 10 λεπτά περισσότερο και να κηρύξω το πέρας τη συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ.